liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύττω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπη στις 5 Φεβρουαρίου του 2009